αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Σας ε, παρακαλώ, Λέδη Άστο, να πάρετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα μεγάλο δυναμικό νέων εξαγωγικών δυνατοτήτων εμφανίζεται στις ασιατικές αγορές που έχουν βεβαίως μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό αλλά και εμπόδια στις εισαγωγές. Ένας τρόπος να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια είναι χρησιμοποιώντας το μοχλό που μας δίνουν οι διαπραγματεύσεις ελεύθερου εμπορίου. Γι' αυτό ζητήσαμε να προχωρήσουμε με νέες συμφωνίες, με οικονομίες κλειδιά της Ασίας. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να δώσουν σε εξαγωγικές δυνατότητες για πολλούς τομείς. Αυτό το πετύχαμε με την Κορία μετά από δύο έντονα χρόνια διαπραγματεύσεων. Είναι η πιο ε, φιλόδοξη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που έχει διαπραγματευτεί ποτέ ε, η Κομισιόν. Τα πλέον εκτήματα από την συμφωνία αυτή είναι οπωσδήποτε υπερημών. Πρώτα απ' όλα, οι ε, παροχής υπηρεσιών θα κερδίσουν πάρα πολλά από αυτή τη συμφωνία στις τηλεπικοινωνίες, στις οικοδομές, στις περιβαλλοντικές υπηρεσίες, θα μπορέσουν δηλαδή να προχωρήσουν σε επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κορέα, στην Κορέα ευκολότερα. Η Κορέα επίσης θα καταργήσει το υψηλό δασμολόγιο. Είναι 35% κατά μέσον όρο. Και τα αγροτικά, οι αγροτικά τους εξαγωγές είναι τα γαλοκτομικά, τα χοιρινά και θα εξασφαλίσουμε και την προστασία των γεωγραφικών προελεύσεων της Ευρώπης. Η, ελεύθερη, ε, η Συμφωνία ελεύθερη εμπορίου, Ελευθέρου Εμπορίου με θα προστατεύσει και τους κατασκευαστές, τους Ευρωπαίους. Θα εξοικονομήσουν 1,2 δις ευρώ σε δασμούς ετήσια. 100 εκατομμύρια την πρώτη μέρα. Οι εξαγωγείς δηλαδή μηχανωμάτων θα εξοικονομήσουν 450 εκατομμύρια ευρώ από την πληρωμή δασμών. Αυτοί που εξάγουν χημικά θα εξοικονομήσουν 150 εκατομμύρια από δασμούς. Η εξαφάνιση των δασμών επίσης θα ενισχύσουν την ε, θέση των εξαγωγέων μας. Οι Κορεάτες, πελάτες, ε, αγοράζουν 25 δις προϊόντα ΕΕ. Σημαίνει ότι η Κορέα είναι πολύ σημαντική αγορά εξαγωγών για μας. Επίσης, η συμφωνία περιλαμβάνει τη διαφάνεια στα αριθμιστικά, καλύτερη προστασία της πνευματικής ε, ιδιοκτησίας και κανόνες για τις ενισχύσεις. Όλα αυτά προς όφελος όλων των κατασκευαστών, των μεταποιητών που πουλάνε προϊόντα στην Κορέα. Βεβαίω υπάρχουν και τα τεχνικά εμπόδια για τα ηλεκτρονικά, τα φαρμακευτικά ε, έχουμε ένα ρυθμιστικό πρότυπο στην Ευρώπη το οποίο εισαγάγαμε σε αυτή τη συμφωνία και έτσι θα ανταποκριθούμε στις απαιτήσει αυτού του κλάδου. Η Κορέα πρέπει να μεταβάλει το, στις εσωτερικές ρυθμιστικές για να συμμορφωθεί ενώ δεν χρειαζόμαστε καμία μεταβολή στην Ευρώπη. Όσον αφορά τώρα ειδικότερα την αυτοκινητοβιομηχανία θα ήθελα να αναφέρω ότι ενδιαφερόμεθα να ενισχύσουμε την πρόσβαση ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στην Κορέα οι εξαγωγής μας είναι η ισχυρότερη εισαγωγή στην κορεατική αγορά. Μπορούν να αναπτυχθούν και άλλο εφόσον θα υποφεληθούν από το συνδυασμό της κατάργησας των δασμών 2.000 ευρώ οικονομία σε δασμούς ενός αυτοκινήτου που στοιχίζει 25. Δηλαδή η συμφωνία περιλαμβάνει πραγματικά ένα σχέδιο κατάργησης δασμών πάρα πολύ φιλόδοξο και πετυχημένο. Τώρα, ένα αυτοκίνητο το οποίο συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα θα θεωρείται ότι συμμορφώνεται και με τα κροατικά πρότυπα, πράγμα που στο παρελθόν ήταν μεγάλο εμπόδιο. Επίσης, υπάρχει ισοτιμία και αντιστοιχεία μεταξύ περιβαλλοντικών ε, ρυθμίσεων μεταξύ Κορέας και, και ακόμη πριν τεθεί η συμφωνία ενισχύ η Κορέα δέχεται ορισμένες μεταβατικές διατάξεις για τα περιβαλλοντικά θέματα που είναι σημαντικά για τους εξαγωγείς και συνεχίζουμε τις συζητήσεις για νέες ρυθμίσεις να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ώστε να μην μπορεί το εμπόριο. Βεβαίως γνωρίζουμε τις ευαισθησίες της βιομηχανίας. Ζητήσαμε μακρά μεταβατική περίοδο για τα μικρά αυτοκίνητα που είναι ευαίσθητα. Οι δασμοί θα καταργηθούν το πέμπτο έτος της συμφωνίας, πράγμα το οποίο δίνει δυνατότητα προσαρμογής. Επίσης υπάρχει σημαντική επένδυση της Κορέας στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Κανόνες προέλευσης τώρα. Αυξήσαμε σε 45% από 40% και έχουμε και διμερή ρήτρα διασφάλισης για δασμούς σε περίπτωση ζημίας της βιομηχανίας. Τώρα Όσον αφορά το drawback για τους δασμούς, δεν είναι τίποτα καινούργιο αυτό, αυτό είναι νόμιμη πολιτική. Η, το drawback των δασμών δεν δίνει σημαντικό πλεονέκτημα ανταγωνισμού για την αυτο, το βιομηχανία μας, διότι έχουμε χαμηλούς δασμούς και τους χαμηλώνουμε περαιτέρω και έχουμε διαπραγματευτεί και ειδική ρήτρα ώστε να σταματήσει τελικά το drawback των δασμών. Υποστηρίζω λοιπόν ότι πραγματικά στηρίξαμε την αυτοκινητοβιομηχανία και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υπηρεσιών μέσω αυτής της συμφωνίας. Αυτό είναι σημαντικό και καταδεικνύει ότι είμαστε επίμονες στην επιδίωξη της θέσης μας κλειδί στις ασιατικές αγορές. Σας ευχαριστώ. Άστον, τώρα έχουμε τους εκπρόσωπους των πολιτικών ομάδων, ο κύριος Κασπάρη του ΕΛΤ πρώτα. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Νότια Κορέα είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμφωνία λοιπόν αυτή ελεύθερων συναλλαγών ε, είναι προς το συμφέρον των εργοδοτών μας και των εργαζομένων μας και κυρία Επίτροπα δεν θέλω να σας συγχαρώ ακόμη σήμερα δεν έχει υπογραφεί άλλωστε αυτή η συμφωνία αλλά αν καταφέρετε στην περίοδο αυτή της κρίσης σε μια τέτοια περίοδο που έχουν καταρρεύσει οι εξαγωγές σε όλο τον κόσμο περισσότερο από ποτέ. Αν καταφέρετε να ολοκληρώσετε αυτό το έργο, θα είναι πραγματικά τεράστια επιτυχία, την οποία και σα την εύχομαι ολόψυχα. Γιατί οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών συχνά είναι πολύ αμφιλεγόμενε και η Νότιος Κορέα είναι μια μεγάλη εξαίρεση όμως και ακούω πολλά θετικά μηνύματα από όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την ε, ηλεκτροχημία, ε, όλε τι υπηρεσίε, Ποτέ δεν έχω ακούσει μόνο θετικές ε, ε, εντυπώσεις και από τον τομέα της γεωργίας μάλιστα. Αυτό είναι πρωτόγνωρο και τα αποτελέσματα είναι ασφαλώς θετικά ακόμα και αν κάποιοι κλάδοι ενδεχομένω να ήθελαν να υπάρχει μεγαλύτερη πρόοδος. Για παράδειγμα, υπάρχουν και μερικές εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα στην κατασκευή οχημάτων, αλλά και πάλι δεν είναι απόλυτα τα πράγματα, γιατί κάποιοι είναι και θετικοί στον κλάδο αυτό. Θα ήταν καλό να αξιοποιήσουμε τον, ε, την ευκαιρία προκειμένου να εξουπετερώσουμε αν θέλετε, ενδεχόμενα αρνητικές πτυχές ε, τις συμφωνίες όπως το Capital Reach Clause, για παράδειγμα, τα περιβαλλοντικά, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και ρήτρε θα πρέπει να μην υπάρξουν παρανοήσεις και πραγματικά να περάσουν όλα αυτά που επιθυμούμε για παράδειγμα, καλύτερη υποπτία. Ελπίζω να τεθεί σε εφαρμογή σύντομα η συμφωνία αυτή και να μπορέσουν να ωφεληθούν οι εργοδότε και οι εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστούμε για όλη την προσπάθεια που έχετε καταβάλει. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά τώρα. Ο κύριος Αρίφλα, ο πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα ε, που ε, ένας ε, συντηρητικός συνάδελφος συμφωνεί με την Επιτροπή αν διευκολύνεται και το δικό μου το έργο ως σοσιαλιστή. Ε, επιτέλους θα δοθούν τώρα απαντήσεις ε, στις πολλές ανησυχίες όσον αφορά τον αντίκτυπο της συμφωνίας αυτής ε, μεταξύ της Κορέας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίκτυπο ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Μιλήσατε, Επίτροπε, για συνένεση. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι εδώ και ορισμένους μήνες ορισμένοι κλάδοι βιομηχανίας, αυτοκινητοβιομηχανία για παράδειγμα και συνδικάτα ευχαριστούν την προσοχή μας για τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας. Και εξακολουθούν και σήμερα ορισμένα ερωτήματα να μην έχουν απαντηθεί λυθεί. Ίσως όμως αποφασίσετε να θυσιάσετε την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία για τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, γιατί συμπεριλαμβάνεται αυτή τη ρήτρα η οποία αποτελεί ε, τεράστιο πλεονέκτημα το οποίο δεν έχει δοθεί ούτε καν στι μεσογειακέ χώρε. Ε, ποια είναι η λογική που ακολουθείτε με τόσο λίγο δεσμευτικού κανόνε ε, ε, για την καταγωγή, με τεράστιε συνέπειε όχι μόνο στην βιομηχανία, αλλά και στην κλωστοφιδουργία. Γιατί να υπάρξει τέτοια στρέβλωση του ανταγωνισμού και κυρίω γιατί να δημιουργηθεί αυτό το προηγούμενο. Απέναντι σε αυτού του κινδύνου αλλά και σε άλλου πολλού που δυστυχώ δεν έχω το χρόνο να του αναφέρω αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ω ε, έσχατο μέσο ε, μία ρήτρα διασφάλιση. Ξέρετε όμω, Επίτροπε, δεν είναι αυτόματη αυτή η ρήτρα. Θα είναι πολύ δύσκολο, να μην σα πω αδύνατο, να ενεργοποιηθεί πριν από πέντε χρόνια. Ε, παίρνω ένα και μόνο παράδειγμα. Εάν η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών θα επιτρέψει 5.000 ε, πιο αυτοκίνητα εξαγωγέ ε, στην Ευρώπη, 6.000 θέσει απασχόληση θα χαθούν. Αντίθετα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τρομερού περιορισμού. Ο καθένα θα εξάγει χίλια, ο κάθε βιομηχανό χίλια αυτοκίνητα με συνολική ποσόστοση 6.000. Πώ θέλετε λοιπόν να προχωρήσουμε προ αυτή τη συμφωνία. Σκέφτεστε περαιτέρω διαπραγματεύσει όσον αφορά ορισμένα φιλεγόμενα σημεία. Είναι αίτημα πολλών κρατών μελών και κυρίω του κλάδου τη αυτοκινητοβιομηχανία. Σκέφτεστε περισσότερη διαφάνεια τέλο και περισσότερη σύνδεση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ε, και εδώ μια αρνητική εικόνα. Ε, ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Για τους φιλελεύθερους, ο κύριος Στοίρ, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς θα ήθελα, κυρία Επίτροπε Άστον, να σας ευχαριστήσω εξ ονόματος της ομάδας του ΑΛΔΕ για την ενημέρωση σήμερα το απόγευμα σε αυτή την ε, συνεδρίαση και στην Ολομέλεια. Τα αποτελέσματα προφανώς ε, αναφορικά με τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών βρίσκονται πριν από την ολοκλήρωση, τους από πλευρά των φιλελευθέρων και από πλευρά FDP. Ο στόχος ε, του δίκαιου εμπορίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα γιατί με την ε, χρηματοπιστωτική κρίση εμφανίστηκαν διάφορες τάσεις προστατευτισμού και αυτές οι τάσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν για το συμφέρον των θέσεων εργασία στην Ευρώπη. Ανακύπτει λοιπόν το ερώτημα του ποια είναι η σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την Νότια Κορέα, γιατί επικεντρωθήκαμε στο γύρο της Ντόχα χωρίς να έχουν όμως επιτευχθεί ε, τελικά αποτελέσματα. Γι' αυτό ερωτώ, λοιπόν, Επιτροπέ Άστον, θεωρείτε ότι με τη σύναψη της συμφωνίας με την Νότια Κορέα γίνεται ένα πρώτο βήμα για περαιτέρω μερή συμφωνίε. και συμφωνείτε ότι μάλλον πιστεύετε ότι πρόκειται για μια, έναν εκτροχιασμό αν θέλετε από το γύρο της Δόχας ή πρόκειται για μια διεύρυνση της πολιτικής ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως γνωρίζετε αυτή η ρήτρα επιστροφής των δασμών για πολλά κράτη-μέλη και για πολλούς κλάδους προκαλεί α προβληματισμό γιατί μπορεί να ενισχύσει τον ανταγωνισμό υπέρ χωρών όπως η Ινδία και η Κίνα. Θεωρείτε ότι αυτές οι αμφιβολίες των κρατών μελών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος, η κυρία Φεγγερέιδο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δήλωση της Επιτρόπου καταδεικνύει ότι Υπάρχουν κλάδοι, οικονομικοί κύκλοι και κλάδοι, οι οποίοι, θέλουν, οι οποίοι πρόκειται να υποφεληθούν από τη συμφωνία αυτή, αλλά υπάρχει και η αντίθετη πλευρά του νομίσματος, κυρία Επίτροπε, την οποία δεν αναφέρατε. Υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, όπως για παράδειγμα η κλωστοφαντουργία και εδώ μιλάμε για θέσεις εργασίας. Και ως εκ τούτου οι κλάδοι αυτοί και οι εργαζόμενοι στις χώρες μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Ότι στην Επιτροπή δηλαδή εξακολουθεί να, η Επιτροπή εξακολουθεί να αγνοεί την ε, άσχημη κατάσταση του κλάδου της κλωστοϊφαντουργίας. Για παράδειγμα, στην χώρα μου επικρατεί μεγάλη ανησυχία. Υπάρχουν είναι πολύ μεγάλες οι ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική η οποία θα προασπιστεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία, ιδιαίτερα την ευρωπαϊκή βιομηχανία ένταση εργασία. και αυτό θα πρέπει να περάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει να υπάρξει πολιτική σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και το καταξή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είναι η παρθενική μου ομιλία αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα περίμενε κανείς να είμαι επαναστάτης βέβαια από εκεί που προέρχομαι, αλλά θα προσπαθήσω να μην σας απογοητεύσω. Συζητούμε συμφωνίες εμπορικές και ειδικότερα με την ε, Νότια Κορέα. Πρόκειται να υπογραφεί φέτος. Επειδή δεν έχουμε και τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας, ε, ε, νομίζουμε ότι υπάρχουν ωφέλη από τη μία πλευρά και από την άλλη, θα ήθελα να κάνω γενικά σχόλια. Εκατό δύο συμφωνίες σαν και αυτοί υπάρχουν. 116 μάλιστα εκτιμάται ότι είναι ο αριθμό. Με τον Καναδά, τη ΣΥΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Νότια Αφρική κτλ. Με την Ευρώπη έχουμε τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Τουρκία και το Λίχτενστάιν. Εμπορικές συμφωνίες έχουμε ακόμη και με χώρες όπως η Ελβετία και η Νορβηγία, χώρες ΕΖΕΣ. Η Συμφωνία ε, της Νορβηγίας προστατεύει και τη γεωργία της και την αλληλεία. Είναι η έκτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά. Τώρα, η Νότια Κορέα, τι θα περιλαμβάνει η συμφωνία. Η Ελβετία είναι καλό παράδειγμα. Υπάρχουν ρυθμίσεις που καταργούν τους δοσμούς, τις ποσοστώσεις για τα γεωρικά και τα βιομηχανικά προϊόντα. Υπάρχουν διατάξεις που επιτρέπουν στους Ελβετούς επικόους να ζουν και να εργάζουν στις χώρες ΕΕΚ και το αντίστροφο. Υπάρχουν διατάξεις να είναι μέλος του Σέγγεν η Ελβετία. Η Ελβετία μπορούν να μπουν στον οργανισμό περιβάλλοντος, ταινιών, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και μπορούν να τύχουν και χωριών για έρευνα, συνεργασία με τις αεροπορικέ γραμμές, για το ασύλο και για τα δικαστικά. Δηλαδή έχουν όλα τα πλεονεκτήματα να είναι μέλη της ΕΕ χωρίς το κόστος. 600 εκατομμύρια πληρώνει για πρόσβαση, αλλά η Ελβετία. Αλλά η ελβετική κυβέρνηση λένε, λέει ότι εξοικονομεί 3,4 δις δηλαδή 2,8 δις καθαρά. 80% των εξαγωγών της Ελβετίας πάνε στην ΕΕ και είναι ο τέταρτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ. Θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να έχουμε ωφέλη χωρίς ρυθμιστικό κόστος, απώλεια καλή κυριαρχίας και πόρων. Ακόμη και ο ιστότοπος... Ναι, με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, πρέπει να σας διακόψω διότι έχουμε ε, συγκεκριμένο χρόνο ομιλίας. Με συγχωρείτε, τι είναι το Blue Card, η διαδικασία Blue Card. Είναι η νέα διαδικασία που κάθε μέλος μπορεί να θέσει ερωτήσεις. Θα ήθελα να τελειώσω όμως, αν μου επιτρέπετε. Μία φράση. Αν δεν συμφωνείτε με τον επόμενο ομιλητή, θα ήθελα να τελειώσω το χρόνο μου ομιλία. Λοιπόν, η Ελβετία μπορεί να αναπτύξει και να διατηρήσει τι ρυθμίσει τη σε άλλου τομεί που διαφεύγουν των διατάξεων, ε, όπω για τα χρηματοπιστωτικά και την αγορά εργασία. Τώρα, και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ήθελε να αποφύγει τις διάφορες ε, ε, οδηγίες που αφορούν το εργασιακό. Και το ερώτημα μου είναι γιατί δεν μπορεί η Βρετανία να έχει μια καλή συμφωνία συνεργασίας με την ΕΕ αντί να είναι μέλος. Είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και έχουμε 40 δις έλλειμμα σε αυτό το ισοζύγιο το εμπορικό με την ΕΕ θα έπρεπε να έχουμε τα ίδια προνόμια με τους Ελβετούς. Θα έπρεπε να είμαστε ένα ανεξάρτητο εμπορικό κράτος όπως η Νορβηγία, η Ελβετία και η Νότια Κορέα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κάμπολ. Ακούσαμε τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και τώρα έχουμε τους άλλους ε, ομιλητές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Πρώτα απ' όλα ε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Στάσινη. Thank ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε, ως ένας από τους συζητητές για, το θέμα της ε, Νότιας Κορέας, ελπίζω να έχουμε μια συμφωνία δίκαιη και ισότιμη που να ε, ωφελεί όλους σε μια κατάσταση win-win. Πρέπει να σα πω ότι η βιομηχανία μα δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη με, με την υφιστάμενη κατάσταση των διαπραγματεύσεων και υπάρχουν ε, ε και κράτη-μέλη τα οποία έχουν τι απόψει και μέλη του Κοινοβουλίου. Ε, πιστεύουν ότι είναι ενισομερή συμφωνία αυτή και ωφελεί ιδιαίτερα την Κορέα. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια για να ε, αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που δημιουργούν τριβέ, μη δεσμολογικά εμπόδια, κανόνε καταγωγή κτλ. Θα μπορούσε να υπάρξει κάποια πρόοδο έτσι ώστε να ικανοποιηθεί περισσότερο η βιομηχανία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με αποτέλεσμα να διατηρηθούν ε, ορισμένα κεκτημένα και από την άλλη ε, να δούμε πώς θα είναι πιο ισότιμη η συμφωνία. Να αντλήσουμε παραδείγματα από άλλες συμφωνίες καθώς και, ε, που, ήδη υπάρχουν και άλλες που έρθουν στο άμεσο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να ωφεληθεί τα μέγιστα από τη συμφωνία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διάφοροι κλάδοι της βιομηχανίας. Πάντα βεβαίω θα υπάρχουν ε, νικητέ ε, και ιτημένοι. Αυτό βρίσκεται στη φύση ε, κάθε διμερού συμφωνία. Αυτά όμω ω προ λεπτομέρειε. Συνολικά όμω θα πρέπει ε, να χαρακτηρίζονται αυτέ οι συμφωνίε από, ε, από, από ισορροπία. Το θέμα τη αυτοκινητοβιομηχανία όμω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο θα υπάρξει προσπάθεια στο τομέα αυτό θα μπορούμε να μιλήσουμε για μια συμφωνία που θα έχει φετικό αντίκτυπο και θα αποτελέσει και προηγούμενο για μελλοντικέ τέτοιε συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σούστα για δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε, σε αυτό το χρονικό διάστημα ε, ε που ε, ε, η Επίτροπος ασκεί τα ε, καθήκοντά τη, είχα την ευκαιρία να εκφράσω το θαυμασμό μου για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντά της. Και βεβαίω πέραν των κοινών πολιτικών πεπιθήσεων και πραγματικά νομίζω ότι οι σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ καλύτερες αυτή τη φορά. Όμως πρέπει να σα πω ότι αυτή τη φορά δεν θα δει δείξω τον ίδιο ενθουσιασμό όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, ενθουσιασμό που έδειξε η Επίτροπος, γιατί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει έρθει εδώ στο Κοινοβούλιο ε, μιλώντας για ορισμένε πρωτοβουλίε ε, και ε, ε, ε, ε, τονίζοντας τα θετικά του σημεία και στη συνέχεια τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως μα είχε πει η Επιτροπή. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή διανύουμε μια πάρα πολύ σημαντική κρίση που προέρχεται και από την απουσία αμοιβαιότητα με τον υπόλοιπο κόσμο. και όχι μόνο σαν αφορά τι αναπτυσσόμενε χώρε, αλλά και όσον αφορά τους νέους πρωταγωνιστές στην, οικονομική, ε, στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Νομίζω λοιπόν ότι πολύ συχνά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ο, ο πρόεδρο τη αλλά και οι Επίτροποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει ποιες πρωτοβουλίε απαιτούνται για να συμβάλλουμε στην ανάκαμψη τη ευρωπαϊκή βιομηχανία. και τη ε, μεταπητική βιομηχανία. Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία, που είναι σωστό, ότι είναι θετική συμφωνία και περιέχει ορισμένα στοιχεία τα οποία είναι θετικά, αλλά φοβάμαι ότι ε, θα έχει ακαδημαϊκή ισχύ χωρί να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Εμεί εξάγουμε 30 δι προ την Κορέα μόλις 20 δις ε, δολαρίων έρχονται με τη μορφή ε, αυτοκινήτων που εξάγονται ε, στην Ευρώπη. Λάβετε υπόψη και τις έμεσες ενισχύσεις με τον τρόπο αυτό θα λάβουν οι Κορεάτες από την Ευρώπη. Και δεν μιλάω για την κλωστοφαντουργία για άλλους τομείς. Εδώ μιλάμε για σαφή έλλειψη ισορροπίας που θα πρέπει να διορθωθεί πριν δώσουμε το πράσινο φω σε μια συμφωνία ελεύθερης συναλλαγών που τιμωρεί την, ε, ε, την αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης που χαρακτηρίζεται από ποιότητα που αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις και που αντιλαμβάνεται ε, τις ε, ανάγκες σύγχρονης οικονομίας. Σας ευχαριστούμε. Να δώσω το λόγο στην κυρία Ροϊτόβα. Ε, Κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, ε, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πολύ καλά αυτά τα θέματα, όπως για παράδειγμα η μείωση του κατοφλίου ε, για, το, για την ε, ε χώρα προέλευσης ε, ή για την ρήτρα αυτή της έκπτωσης. Όλα αυτά θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρώπη. Σήμερα, κοιτάξτε, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των ασιατικών προϊόντων, όπου το, το εργατικό δυναμικό είναι ιδιαίτερα φθηνό, αλλά δεν υπάρχουν κοινωνικοί κανόνες και κανόνες προστασία των εργαζομένων. Λοιπόν, κοιτάξτε, ε, η βελτίωση των κανόνων αυτών θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο των ε, διαπραγματεύσεων αυτών. Ε, να λοιπόν, έχω συγκεκριμένε ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε συνειδητοποιήσει τον αρνητικό αντίκτυπο τη συμφωνία στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, στην απασχόληση. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι υπάρχει ένα ολέθριο προηγούμενο το οποίο θα μπορούσε να επιδράσει, ε, θα δημιουργηθεί λοιπόν ολέθριο προηγούμενο που θα επιδράσει και στις μελλοντικέ ε, ε, συμφωνίες. Θα λάβει υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Επιφυλάξης των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Ήδη όμως ο τύπος στην Κορέα γιορτάζει και θρεμολογεί, ενώ δεν έχει συζητηθεί ακόμα συμφωνία από το Σώμα των Επιτρόπων. Είναι έτοιμη η Επιτροπή ε, να επανεξετάσει ενδεχομένως το ζήτημα και να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους ή ε, θα ε, ασκηθεί πίεση ή θα ασκήσει πίεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Κορέα να σεβαστεί τις διεθνείς δεσμεύσεις. Ελπίζω τελικά να θριαμβεύσει λογική. Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι ανησυχώ με τον τόνο αυτής με αυτή της με εξαίρεση τη συμβολή του Ντάνιελ Κασπάρη. Είναι αρνητικά τα σχόλια. Ήμουνα εισηγητή στην έκθεση και ζητήσαμε από την Κομισιόν να προχωρήσει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, να πετύχει ορισμένα αποτελέσματα και νομίζω ότι η Κομισιόν πετύχει ακριβώς αυτά τα οποία ζητήσαμε. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον επικεφαλής ε, της ομάδας διαπραγμάτευσης για τον τρόπο με τον οποίο καταφέρανε να καταλήξουν σε αυτή τη συμφωνία. Βεβαίως υπάρχουν πάντοτε νικητές και ηττημένοι αλλά το γενικό αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας είναι μεγάλοι νικητές στην Ευρώπη, αλλά και στην Κορέα. Και έτσι προωθείται το εμπόριο. Και στη σημερινή κρίση οτιδήποτε μεταδίδει ένα θετικό μήνυμα από δύο αγορές όσο, σημαντικές όσο η Κορέα και η ΕΕ ένα θετικό μήνυμα λοιπόν είναι πάντοτε μεγάλο πλεονέκτημα. Το Συμβούλιο δεν μπορεί Αν δεν προχωρήσει λοιπόν αυτή ε, η συμφωνία στο Συμβούλιο των Υπουργών, θα έπρεπε να πούμε στη Γενική Διεύθυνση να σταματήσει να διαπραγματεύεται. Διότι αν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την Κορέα, ξεχάστε τις χώρες του Κόλτου και, και την Τόχα. Ειλικρινά είναι μια σημαντική συμφωνία με την Κορέα. Η Ευρώπη έχει πετύχει τους στρατηγικούς στόχους της. Ας περάσουμε ένα θετικό μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο ότι είναι επιχειρηματική η Ευρώπη και διατηρεί τις αγορές της ανοιχτές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε το λόγο τώρα μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ο κύριος Κέλλη. Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Βρήκα τη συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα και εκπαιδευτική. Όταν πρωτομίλησε η Lady Άστον, σκέφτηκα ότι είναι πολύ καλή η συμφωνία γιατί είναι αναρωτιόμουν και τι κερδίζει η Κορέα. Αλλά μετά τους διάφορους ομιλητές ε, έχω καταλήξει στην αντίθετη, στο αντίθετο συμπέρασμα. Ελπίζω λοιπόν ότι τα σχόλια των ομιλητών θα απαντηθούν πολύ συγκεκριμένα από τη λέει Διάστον στην απάντησή της. Επίσης θα μπορούσε να μας πει αν υπάρχουν άλλες διαπραγματεύσεις που προωθούνται αυτή τη στιγμή με συγκεκριμένες ασιατικές χώρες. Πόσο έχουν προοδεύσει ενδεχομένες τέτοιες διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη, ο κύριος Μπάτον. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω τον ισχυρισμό του συναδέλφου Κάρμερ Μπάνεμαν. Το 2006 η ελβετική κυβέρνηση ε, συνέταξε μία έκθεση σε σχέση με όλες τις σχέσεις με την ΕΕ. Δηλαδή εξέτασε τι θα στήχιζε να γίνουν πλήρη μέλη. Έξι φορές τις σημερινέ τους δαπάνες θα στήχιζε το να γίνουν μέλη και οι Ελβετία, επειδή είναι Ελβετοί, αποφάσισαν ότι καλύτερα να μην μπουν στην ΕΕ. Αν αυτό ισχύει λοιπόν για τους Ελβετούς, σίγουρα ισχύει και για τους Βρετανούς. Μακάρι η κυβέρνησή μας να είχε μια τέτοια ρεαλιστική αντιμετώπιση της οικονομίας όπως οι Ελβετοί. Θα φεύγαμε κι εμείς όπως δεν μπαίνουν οι Ελβετοί. Διαδικαστικό ο κύριος Μάρτιν ζητά. Είσαστε πολύ υπομονητικός πρόεδρος κύριε πρόεδρε, αλλά είναι σαφές ότι βάσει του Catch the Eye πρέπει να παρεμβαίνει κανείς στο θέμα. Δεν είχε, το σχόλιο αυτό που έκανε ο κύριος δεν έχει καμία σχέση με την Κορέα για την εμπορική συμφωνία. Ήταν άσχετο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ισάια τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Μόρτιν στην παρέμβασή του υπενθύμησε ότι στην κατάσταση κρίση που αντιμετωπίζουμε είναι πολύ σημαντικό να οδηγηθούμε σε συμφωνίε που θα υποκινήσουν τι εμπορικέ συναλλαγέ, θα καταργήσουν τα εμπόδια στο εμπόριο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σήμερα είχαμε μια πολύ σημαντική συζήτηση για την κρίση της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Ε, αναφερόμαστε και στην κρίση της φαντουργίας και στις απολύσεις της μαζικές που εμφανίζονται στην Ισπανία και στην Πορτογαλία σε ορισμένους κλάδους. Κυρία Επίτροπε, σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις απώλειες εργασίας, να δοθεί μία απάντηση από την Κομισιόν. Βεβαίως χρειάζεται το ελεύθερο εμπόδιο αλλά τι γίνεται με την απασχόληση στους παραδοσιακούς κλάδους της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Έχετε πολλά, πολλές ερωτήσεις να απαντήσετε. Έχετε το λόγο, κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι η συζήτηση δεν ε, μου προκάλεσε έκπληξη, γιατί οι ανησυχίες που έθιξαν οι συνάδελφοι όντως ε, αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια των μηνών και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον David Martin για τη δουλειά που έκανε στην Επιτροπή. Είναι πολύ σημαντικό και αναγνωρίζω πόσο συνεργάστηκε μαζί μου η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου τους προηγούμενους μήνες και φυσικά συνειδητοποιώ ότι συνάδελφοι που δεν έχουν εξετάσει τις λεπτομέρειες της συμφωνίας μπορεί να έχουν ανησυχίες. Θα προσπαθήσω να τις καθησυχάσω, αλλά πιο σημαντικό θα προσπαθήσω να διασφαλίσω ότι θα σας δώσουμε όλο και πιο πολλές λεπτομέρειες, γιατί θα πρέπει, και είναι σημαντικό αυτό, να κοιτάξουμε ποια είναι τα γεγονότα. Ποια είναι η πραγματικότητα. Να πω λίγα γενικά πράγματα για τη γενική προσέγγιση καταρχάς. Η συμφωνία αυτή ξεκίνησε προκειμένου να επιτευχθεί ό,τι καλύτερο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία συμπεριλαμβανομένης και της βιομηχανίας ε, της Βρετανικής, να πω στους συναδέλφους της UKIP. Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης, απόλυτα θεωρώ, να προχωρήσει η συμφωνία αυτή. Ή δεν θα στεκόμουν εδώ ενώπιόν σας να προτείνω την ολοκληρώση της συμφωνίας αυτής. Ωστόσο, ήταν σαφής η προσέγγιση που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, όπως τονίστηκε, έτυχε της υποστηρίξεις και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Αυτός ήταν ο τρόπος που ακολουθήσαμε και οι συνάδελφοί μου ελπίζω να εκτιμήσουν αυτό που θα πω. Δεν σκοπεύω να θυσιάσω οποιαδήποτε βιομηχανία. Αλλά αν θέλουμε μια σοβαρή συμφωνία, προφανώς θα πρέπει να γνωρίσουμε ότι πρόκειται για μια συμφωνία η οποία θα θέλει και τις δύο πλευρές. Αν θέλουμε να υπάρχουν τέτοιες εμπορικές συμφωνίες, το εμπόριο θα είναι η κινητήριος δύναμη που θα μας βγάλει από την κρίση. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν σοβαρές, σκληρές διαπραγματεύσεις και με τους κλάδους και με τις χώρες τις οποίες, οι οποίες μας ενδιαφέρουν ως προς τη σύναψη συμφωνιών. Ή δάλλως, να κάνουμε συμφωνίες με χώρες όλη μέρα που δεν μας ενδιαφέρουν. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν πραγματικά οι αγορές μας, οι αγορές τους. Η Κορέα αποτελεί μια σημαντική αγορά με σημαντικές ευκαιρίες για τα χημικά, τη φαρμακοβιομηχανία και άλλες βιομηχανίες. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε τη σημασία της δράσης αυτής. Αν θέλετε, τονίζω, αν θέλετε σοβαρές εμπορικές σχέσεις Είμαστε οικονομική υπερδύναμη. Δεν, διαφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα με τους συναδέλφους από τον Εμένε Βασίλειο όταν μιλούν για την Ελβετία και προσπαθούν να εξισώσουν, αν θέλετε, τις σχέσεις που προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε με την Νότια Κορέα. Αυτό εννοείται, γιατί δεν καταλαβαίνω. Πρόκειται για σοβαρές διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη σοβαρού αποτελέσματος. Και Γνωρίζω τις λεπτομέρειες, ελπίζω να τις κοιτάξουν και οι συνάδελφοι υπό το ίδιο πνεύμα. Για την αυτοκινητοβιομηχανία, ε, εξ αρχής είχαμε ένα κατάλογο στόχων, γιατί ειλικρινά ανησυχούσε ο κλάδος προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή η αγορά στην ε, Κορέα. Για την κλωστοϊφαντουργία, είμαι βέβαιη ότι δεν έχουμε πολλά για να ανησυχήσουμε οι δικλείδες όντως θα διασφαλίσουν, θα διατηρήσουμε τις ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας. Δεν ε, έχω συμφέρον να κλείσουν ευρωπαϊκοί κλάδοι να καταστραφούν θέσεις εργασίας και όλοι όσοι πιστεύουν ότι έχουν αποτεκτικά στοιχεία παρακαλώ να μου τα διαβιβάσουν γιατί άλλο οι εντυπώσεις και άλλο η πραγματικότητα και θα πρέπει να περάσουμε από την ρητορία αν θέλετε στην πραγματικότητα πλέον. Αυτό που έχουμε ενώπιόν μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους βιομηχανικούς κλάδους. Για το duty drawback το θέμα είναι πολύ απλό θεωρώ γιατί έχει σχεδιαστεί για να προλάβει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Το θέμα είναι, είναι ο μοναδικός τρόπος για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό ή υπάρχουν και άλλοι τρόποι που λύνουν εξίσου το πρόβλημα και μας ε, οδηγούν σε μια καλύτερη εμπορική συμφωνία. Να τους ερευνήσω αν υπάρχουν οι τρόποι αυτοί, αλλά το ίδιο πρόβλημα θα επιδιώκω να λύσω. Και πιστεύω ότι οι μηχανισμοί που έχουμε εφαρμόσει ακριβώς αυτό κάνουν. Δεν είναι απλά ένα στοιχείο το οποίο το έχουμε καθιερώσει και το έχουμε ιερό αν θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε επιλύσει το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο. Δεν πρόκειται λοιπόν να απολογηθώ πολιτικά, οικονομικά ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο ενώπιον του Κοινοβουλίου για το γεγονός ότι επένδυσα στις ε, διαπραγματεύσεις για αυτή την σημαντική εμπορική συμφωνία. Δεν απολογούμε καθόλου και δεν απολογούμε καθόλου για το ότι προτείνω στο Κοινοβούλιο αυτό, αυτό που θεωρώ ότι είναι μια σύγχρονη και σοβαρή εμπορική συμφωνία για μια τεράστια σημασία οικονομία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα όταν απολογούμε σε μια εποχή οικονομικής κρίσης γιατί αν, υπήρχε, υπάρχει μια εποχή όπου είναι ακόμα πιο σημαντική η δική μου αρμοδιότητα για, σε ό,τι αφορά τις θέσεις εργασίας και τη βιομηχανία νομίζω ότι ε, αυτή είναι, πιο σημαντικός ε, αυτή είναι η πιο σημαντική εποχή και καλώ τους συναδέλφους να κοιτάξουν την πραγματικότητα. Θα υπόκειστε και στις επιρροές του λόμπι, όπως και εγώ. Αλλά ειλικρινά πιστεύω ότι έχουμε πετύχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα το οποίο θα υποφελήσει πάρα πολύ την οικονομία της Ευρώπης. Αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος μας, αυτό και πετυχαίνουμε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Έληξε και η συζήτηση λοιπόν για το θέμα αυτό και τώρα έχουμε ακόμη ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη, η προφορική ερώτηση, η επιπτώση της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης για τις αναπτυσσόμενες χώρες και την αναπτυξιακή συνεργασία. Και το λόγο, μάλλον να καλέσω τον κύριο Ντεχούχτ να καθίσει στη θέση του και παραλληλού να δώσω στην κυρία Τζολί τον λόγο. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριοι Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,